suis euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ξαναλέει πρόεδρος. Ξανακαθίστε. Ξαναλέει. Συνεχίζεται η συνεδρίασή μας. Έχουμε καθυστέρηση λίγο και θα πρέπει να ζητήσουμε ειλικρινά, ειλικρινά να μας συγχωρήσει ο κύριος Γκάρκοφ ε, και θα του δώσουμε σε λίγο το λόγο. Και θα πρέπει να δούμε το, τι έγινε το εξή. Ενώ υπάρχει στην Ολομέλη ζήτηση για το Λίζα, έχουμε και εδώ τον Διευθυντή. Οπότε κάποιοι συνάδελφοι οφείλουν να βρίσκονται στην Ολομέλη, στο ημικύκλο δηλαδή. Οπότε έχουμε, α πούμε, την κυρία Κινίτσε που πρέπει να πάει. Αλλά πριν σα δώσω το λόγο, θα πρέπει να σας πω ότι 21 Τρίτο το πρωί έχουμε συνεδρίαση και το απόγευμα 2.30 με 6.30 και στις 9 Μαρτίου το πρωί στις Βρυξέλλες. Αυτά προς ενημέρωση. Στις 22 Μαρτίου το πρωί και στις 21 Μαρτίου όλη την ημέρα. Και τώρα, ο κύριος Γκάρκοφ είναι ο εξωτερικός διευθυντής του Λίζα. Όλοι θα γνωρίζετε ότι πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την επιχειρησιακή διαχείριση των συστημάτων πληροφόρησης. Και συγκεκριμένα έχει αναλάβει το σύστημα SIS, το σύστημα πληροφοριών του Schengen, αλλά και το VIS, αλλά και το Eurodac για όλα τα προβλήματα, για όλα τα κενά, για τις, ε, την, ανταλλαγή των πληροφοριών στην πράξη. Αυτά που τώρα είναι όλα στο θεματολόγιο της Ένωσης. Ε, γι' αυτό και εμείς σας καλέσαμε να έρθετε να λύσετε τις απορίες των συναδέλφων. Ε, δηλαδή η εντολή μας είναι στενά στεδεμένη με αυτά τα επιχειρησιακά θέματα που είναι στην αρμοδιότητά σας και σχετίζονται βέβαια και με την υπηρεσία Λίζα. Επίσης, αφού κάνετε την ε, εισήγησή σας, εάν θέλετε και πώς να μην θέλετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Τις τυχόν ερωτήσεις των συναδελφών ε, που θα απευθύνονται σας. Έχετε τον λόγο, κυρία Γκάρκαφ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής σας και ευχαριστώ για αυτή την ε, ευκαιρία να σας παρουσιάσω τι μπορεί να μας προσφέρουν οι νέες τεχνολογικές λύσεις για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Παρακολουθήσα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την προηγούμενη συζήτηση και ξέρω ότι η Ευρώπη σήμερα αντιμετωπίζει νέες απειλές. Θέλει να παραμείνει από τη μία ανοιχτή στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά από την άλλη θέλει να είναι και ασφαλής. Οι πολίτες μας έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν ε, ασφαλείς και να αισθάνονται ασφάλεια στις χώρες τους, στα σπίτια τους. Γι' αυτό η ασφάλεια των πολιτών είναι μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις των τελευταίων ετών, μια πρόσφατη μελέτη του Ευρωβαρομέτρου δείχνει ότι 95% των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η τρομοκρατία είναι μια νέα απειλή. Γι' αυτό η καταπολέμησή της θα πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας. Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια δείχνει ότι μια από τις τρεις προτεραιότητες επίσης είναι η τρομοκρατία και η καταπολέμησή της και είναι ένας χώρος όπου μπορεί να κάνει τη διαφορά η Ευρώπη να είναι πρωτοποριακή στη δράση της. Σήμερα βλέπουμε ε, και είμαστε μάρτυρες ενός φαινόμενο. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας από τις δυνάμεις ασφαλείας ε, συνολικά βασίζεται στις πληροφορίες, τα δεδομένα, τις πληροφορίες και την ανταλλαγή τους. Γι' αυτό τα συστήματα για τα οποία είμαι υπεύθυνο και για τα οποία θέλω να σας μιλήσω σήμερα θα παίζουν και στο μέλλον ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη μιας εύστοχης και αποτελεσματικής απάντησης στις τρομοκρατικές απειλές που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη να ξεκινήσω με κάποια προφανή στοιχεία που είναι προφανή και από την προηγούμενη συζήτηση. Το σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών Schengen είναι σήμερα το πιο δυνατό ε, σύστημα πληροφορική τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για την ε, εσωτερική μα προστασία και χρησιμοποιείται από τι διοκτικέ και δικαστικέ αρχέ για να εντοπίζουμε σοβαρό οργανωμένο έγκλημα μεταξύ των οποίων και τρομοκρατία. Ε, κάνει ελέγχου σε ανθρώπους και εντοπίζει απειλές κατά τη ασφάλεια. Το 2014 το Συμβούλιο ζήτησε συγκεκριμένε δράσει από την Επιτροπή για να ενισχύσει και να ενδυναμώσει την απόκριση στην τρομοκρατία, στην απειλή της τρομοκρατίας και αυτό άρχισε να γίνεται εν γέννη πράξη το 2015. Έκτοτε αυτό που είδαμε είναι μια τάση να χρησιμοποιείται ακόμη περισσότερο το σύστημα Σέγγεν. Το 2016 είχαμε πάνω από 4 δις, 4 δις ε, αναζητήσεις στο σύστημα. Τα προσωρινά δεδομένα για το 2017 δείχνουν ότι μπορούμε να περιμένουμε 25% περισσότερες αναζητήσεις. Αυτό σημαίνει ότι το ΣΥΣ2 την χάνει αναγνώρισης από την κοινότητα των διοκτικών αρχών στην Ευρώπη ως το πιο σημαντικό ε, εργαλείο και πιο σημαντική πλατφόρμα για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών. Και αυτό αυτό σε σχέση με την καταπολέμηση τρομοκρατικών ε, επιθέσεων. Ε, τώρα, για το άρθρο 36 που αναφέρθηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές, το τέλος του 2017 σηματοδοτεί 30% αύξηση της ε, αποθήκευσης των δεδομένων στο σύστημα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2016, δηλαδή δύο χρόνια πληροφοριών βάσει του άρθρου 36 στο σύστημα ε, δύο χρόνια δεδομένων διπλασιασμός των πληροφοριών. Αυτό δείχνει τη διεύρυνση του συστήματος και τη σημασία που αποδίδουν οι δικτικές αρχές της Ευρώπης στο όλο εγχείρημα. Αυτό δείχνει και τη σημασία της ε, χρήσης του συστήματος. 20% αύξηση των ε, αναζητήσεων δίνει και περισσότερα αποτελέσματα το σύστημα και στο πλαίσιο των συστηματικών ελέγχων των ε, όσων φτάνουν στα εξωτερικά σύνορα και άρχισαν να ισχύουν επισήμω από το 2017, το ΣΥΣ2 δίνει μια δυνατότητα ε, πλατφόρμας με εργαλεία για τους συνοροφύλακες για την καλύτερη διεξαγωγή των καθηκόντων τους για να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις νέες προκλήσεις και δυσκολίες ε, με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότητα στους ε, τακτικούς ελέγχους. Δεν... χωρίς να απαιτείται η βελτίωση των επιδόσεων των εθνικών συστημάτων. Είναι σημαντικό το σύστημα σήμερα να παραμείνει ε, λειτουργικό και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, άμεσα τώρα που το χρειαζόμαστε, αλλά και στο μέλλον. Οι τρομοκράτε ε, μεταβάλλουν τη δράση του. Τα ίδια πρέπει να προσαρμόζονται κατά συστήματα, ιδίω το συστήμα, ω βασικό εργαλείο για να ε, στηρίξει τι προσπάθειε των διοικητικών αρχών στην Ευρώπη και να δίνουν συνεχώ τι κατάλληλε αποκρίσει. Γι' αυτό το πακέτο συστείο έχει κάποιε τεχνικέ και λειτουργικέ ε, βελτιώσει ω προ το σύστημα και τη βασική του λειτουργία. Και αυτή τη στιγμή είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων αυτή η τροποποίηση. Ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα υλοποιηθεί και θα δώσει στον οργανισμό την δυνατότητα να εργαστεί καλύτερα και να δώσει στις διοκτικές αρχές της Ευρώπης την ευκαιρία για πολύ καλές επιδόσεις. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό για το σύστημα είναι ότι σύντομα το ΣΥΣ 2 από τις 6 Μαρτίου δηλαδή θα έχει αναβαθμισμένες δυνατότητες. Θα υπάρχουν τα τόσο σημαντικά βιομετρικά δεδομένα που επιτρέπουν υψηλές επιδόσεις και στι διοκτικέ αρχέ να έχουν ένα προηγμένο εργαλείο για τη δουλειά του. Τα άλλα δύο συστήματα για τα οποία είμαι υπεύθυνο συμβαίνουν και αυτά αμέσω στην ε, καταπολέμηση τη τρομοκρατία, ιδίω το ΒΙΣ. Το ΒΙΣ είναι ένα προηγμένο εργαλείο για το screening ε, των θεωρήσεων. Αυτό από τις υπεύθυνε κεντρικές αρχές αλλά και από τις αρχές ελέγχου των συνόρων με το συστείο. Το ίδιο και για το Eurodac. Από το 2015 είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων και να ε, σας πληροφορήσω ότι από τις 22 Ιουνίου 2017 η Ευρωπόλ είναι συνδεδεμένη στο Eurodac και μπορεί να το αξιοποιήσει για τις ερευνές της. Πάντως, για το Eurodax ισχύουν οι, δύο, οι ίδιες αρχές όπως για το SIS2. Το σύστημα πρέπει να γίνει στεγανό, για, να προσδεθεί για το μέλλον και να προσφέρει τις δυνατότητες στις διοκτικές αρχές, τις αρχές επιβολής του νόμου γενικότερα. Το Eurodac, ως προς τις πληροφορίες του, με τις προσαρμογές του θα παρέχει δύο νέες δυνατότητες. Πρώτα απ' όλα εξελιγμένα εργαλεία για καταλληλότερες αποκρίσεις της μεταναστευτικής πίεση βάσει της μεταρρύθμισης του Δουβλίνου, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Δουβλίνου και μετά νέε δυνατότητες στο σύστημα. Αλφαμετρικά δεδομένα, βιομετρικά, αλφαριθμητικά δεδομένα, ε, βιομετρικά, σημαντικά για τις κοινότητες των διοκτικών αρχών, για να μπορούν να εκτελέσουν καλύτερα τα καθήκοντά τους. Και πάλι, Ελπίζω ότι ο νέος κανονισμός Eurodac θα ε, μεταφραστεί και σε νομοθετική πράξη. Πάντως, ως προς τα νέα συστήματα, ως προς το τωρινό μάλλον σύστημα, τα χρειαζόμαστε και στο μέλλον. Είναι γνωστό ότι το αρχιτεκτόνημα ανταλλαγής πληροφοριών όπου είχε κάποια κενά η Ευρώπη, πρέπει να συμπληρωθεί. Θα είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε σωστή υλοποίηση των νέων συστημάτων που σύντομα έρχονται. Πρώτα απ' όλα το NCRIV system, ε, το σύστημα που ήδη επεξεργαζόμαστε σε πλωτική φάση μετά τη θέση σε ισχύ ε, του κανονισμού στις 29 Δεκεμβρίου του περασμένου έτου, Εδώ δυνατότητα, έχουμε δυνατότητα ανείχνευσης πλαστών εγγράφων, ταυτοτήτων και ταυτοποίησης και αυτό με τη συμμετοχή των αρχών ελέγχου στα σύνορα και των αρχών ταυτοποίησης Επίση για του υπηκόου των χωρών με τρομοκρατικέ προθέσει. Δεν θα μπορούν πλέον ε, χωρί ε, ταυτοποίηση να περάσουν τα σύνορα και θα συμβάλλει αυτό την εσωτερική προστασία της Ευρώπης. Το έτιας θα είναι ένα άλλο σύστημα που θα συμβάλλει περαιτέρω στην εσωτερική ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας καθώς θα βοηθά να εντοπίσουμε τους ε, επικόστητων των χωρών που εξαιρούνται τις υποχρεώσει θεώρηση και να γίνεται ένας έλεγχο ασφάλεια προτού περάσουν τα σύνορα. Έτσι, οι αστυνομικοί και οι συνοριοφύλακες θα είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις πιο εμπεριστατωμένε. Πάντως, σημαντικό είναι να αναφέρω και αυτό στο πλαίσιο και της προηγούμενη συζήτηση που είχατε, ότι τα συστήματα και οι πληροφορίε που ε, χρησιμοποιούνταν απομονωμένα σε σε ξεχωριστά τμήματα ε, θα πρέπει τώρα να συνδυαστούν. Γι' αυτό θα αλλάξει ο σχετικό κανονισμό καθώ και τα όσα προβλέπονται για την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των δεδομένων για την εσωτερική ασφάλεια και την καταπολέμηση τη θερμοκρατία. Διότι πρέπει να διασφαλίσουμε και να προσφέρουμε πιο εξελιγμένα εργαλεία στι εθνικέ αρχέ και του τελικού χρήστε. Για να έχουν τι απαραίτητε πληροφορίε στην κατάλληλη στιγμή και με και στην κατάλληλη ποσότητα για να μπορούν να λαμβάνουν μια τεκμηριωμένη απόφαση. Δεν θέλουμε ε, διωγγωμένη παρουσία δεδομένων ούτε να εμποδίσουμε την καλή διεξαγωγή των καθηκόνων του. Χρειαζόμαστε τι κατάλληλε πληροφορίε στην κατάλληλη στιγμή. Είναι λοιπόν ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του ευρύτερου συστήματος πληροφοριών σε ευρωπαϊκή κλίμακα και όσα προσφέρονται στις αρχές ε, δίωξης και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Και δύο λόγια για την ε, διαλογικότητα και το πώς θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Υπάρχουν τέσσερα σημεία στην ε, ανάλογη πρόταση το κοινό αποθετήριο και ο ε, ταυτότητα. ταυτότητας. Δεν θα μπορούν πια οι υποπτοί να έχουν πολλαπλές ταυτότητες. Για την ε, επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά, ε, ο συγκεκριμένο άνθρωπος είχε 14 ταυτότητες στην Γερμανία και ίσως σε άλλες ευρωπαϊκές ε, δεδομένων. Με το κοινό αποθετήριο δεν θα είναι πλέον αυτό δυνατό. Διότι όλες οι ταυτότητες ε, με τα παραμετρικά δεδομένα θα συνδέονται με το ίδιο πρόσωπο. Οπότε οι εθνικές και οι ευρωπαϊκές αρχές θα είναι σε θέση να λάβουν τα και πιο εμπεριστατωμένε αποφάσει. Οι κοινέ τα κοινά βιομετρικά δεδομένα με το ανάλογο πόρταλ για αναζήτηση θα επιτρέπει στου τελικούς χρήστες να έχουν κατάλληλη πρόσβαση στα δεδομένα με πλήρη σεβασμό των κανόνων περί προστασίας των δεδομένων. Βελτιωμένος λοιπόν τρόπος για να μπορούν οι διοκτικές αρχές να, ε, και οι αρχές ασύλου να υποφελούνται από αυτά. Επίσης για τη διαλογικότητα θα ε, διευκολύνει και θα συμβάλλει στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κατών μελών και θα έπρεπε να είναι σαφές ότι τα νέα συστήματα και οι υποδομές θα χρειαστούν αλλαγές στο προσεχές μέλλον λόγω της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και ευγενικά να σας θυμίσω ότι η Λίζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η EU Λίζα, θα ε, φροντίσει να παρακολουθεί τα συστήματα αυτά και την εξέλιξή του για το πώ χρησιμοποιούνται από τους κατελικού χρήστε. Οι δυνατότητε και οι λειτουργίες τους, λόγω χάρη, για την περίπτωση των ξένων μαχητών. Άρθρο 36, ε, αρχέ του 2015, το πρόγραμμα δράσης για την ποιότητα των δεδομένων, όπου είμαστε συντονιστές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαντικό στοιχείο πολιτική για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων και την ανάπτυξη της απαραίτητης απόκρισης στις διάφορες απειλές. Αρμοδιότητα και αποστολή της, ε, του οργανισμού είναι να παρακολουθεί τις ε, απειλές τεχνολογίες και να προσαρμόζεται σε και να είναι η Ευρώπη ασφαλέστερη. Θέλουμε να είμαστε ένα ε, βασικός παράγοντας για την προστασία της ασφάλειας στην Ευρώπη. Να είστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τα συστήματα και τις υπηρεσίες μα εργαλεία που είναι ζωτική σημασία για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και την εσωτερική ασφάλεια τη Ευρώπη. Θα φροντίσουμε να καλύπτουν τι ανάγκε σα και τη ζήτηση που ενδεχομένω θα αναπτυχθεί στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκάρκοφ για την παρουσίαση αυτή και κυρίω ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ που είναι οι ελπίδες που έχουμε να αποθέσει στο σύστημα ε, διαλειτουργικότητας που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση. Να έχουμε ένα ποιοτικό άλμα ως προς την ιχνηλασιμότητα και την πρόληψη των τρομοκρατικών επιθέσεων. Όλα αυτά είναι επίκαιρα στην Ευρώπη αλλά και στα νομοθετικά κείμενα. Θα δώσω το λόγο στου συναδέλφου. Ο Γερούν Λέναρτ ζήτησε το λόγο. Μετά. Ο Νούνο Μέλο. Άλλος. Εγώ ζήτησα πρώτος, λέει, κύριος Μέλο, χωρίς μικροφόν. Yes. Ε, yes, because ε, ε, nous suivons une sorte de... Κοιτάξτε, έχουμε μια σειρά ιεραρχία εδώ στην Επιτροπή ο Γιώργο Λέναρς. Για ένα λεπτό. Ένα λεπτό ολόκληρο. Καλά. Πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας και για ε, τη φιλοξενία του ε, οργανισμού που επανειλημμένα είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε και με την Επιτροπή Λιμπέλα και προσωπικά σε επίσκεψή μου. Μιλήσατε για την πρόταση διαλειτουργικότητας. Όλοι στο Κοινοβούλιο προσβλέπουν ε, να εργαστούν για αυτό το θέμα εσείς, ο οργανισμός σας, πώς σκέφτεστε να τα αντιμετωπίσετε όλα αυτά. Έχουμε το Eurodac, το SIS, το ES, ε, ενημερώνονται πολλά συστήματα, όχι λόγω της νέας πρότασης μόνο, αλλά γιατί χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο. Και τώρα θα εργαστούμε για την διαλειτουργικότητα. Εδώ είμαστε κοινοβούλιο και όλοι έχουμε οράματα και όνειρα να βελτιώσουμε όσο γίνεται περισσότερο το σύστημα. Με την νέα εντολή βέβαια εσείς πώς βλέπετε τη δουλειά σας και τις δυνατότητές σας να ανταποκρίνονται σε όλα αυτά που ζητάμε να κάνετε. Έχετε αρκετούς πόρους και ανθρωπίνους και, και χρήματα και δυνατότητες για να κάνετε τη δουλειά που ζητάμε από εσάς να κάνετε. Merci, uh, σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Την επόμενη τριετία με πενταετία θα υπάρξουν πολλές πρωτοβουλίες για τις οποίες θα είμαστε αρμόδιοι. Μία από αυτές είναι η διαλειτουργικότητα, αλλά υπάρχουν πολλά. Η ε, αναδιατύπωση του ΣΥΣ2, το σύστημα ε, των θεωρήσεων και πολλά ακόμα. Και προφανώς ε, αυξάνονται πάντα ε, οι προσδοκίες ε, προς εμάς και είναι και μεγάλη πρόκληση. Πολύ σωστά το αναφέρατε. Τι δυνατότητες έχουμε να ανταποκριθούμε και τι πόρους. Για την πενταετία, πενταετία που υπάρχει, πρέπει να σας πω ότι δεν αυξήθηκαν οι υπάλληλοι παρά το γεγονός ότι αυξήθηκαν τα καθήκοντα και η συνεισφορά προς τα κράτη-μέλη και συνεχώς αυξάνονται. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα τώρα να ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα και μάλιστα τα θεσμικά άργονα που είναι αρμόδια για την ε, υπόθεση των πόρων να κοιτάξουν και το γιο Λίζα και να μας δώσουν τους απαραίτητους πόρους για να κάνουμε τη δουλειά μας, αυτό που περιμένετε από εμά. Όταν μιλώ για πόρους, αυτό αφορά δύο ε, πράγματα. Δεν είναι τίποτα καινούριο, αλλά χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας εδώ στο Στρασβούργο το επιχειρησιακό μας κέντρο δεν επαρκεί. Πρέπει να μεγαλώσει ε, και περαιτέρω τον όσο κάνουμε τώρα. και χρειαζόμαστε υποστήριξη από το Κοινοβούλιο, φυσικά και από το Συμβούλιο, ε, που είναι αρμόδιες δημοσιονομικές αρχές. Το δεύτερο και σημαντικότερο βέβαια, εκτός από τα τεχνικά, είναι οι ανθρώπινοι πόροι θα ε, χρειαστούμε γενναία ενίσχυση σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων. Ξέρω ότι πολλές από τις νομοθετικές προτάσεις που καταθέτεται προβλέπουν επιπλέον πόρους, αλλά για ένα ειδικό σκοπό. Για να διατηρηθεί όμως η λειτουργική και επιχειρησιακή δυνατότητά μας και να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε, χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους για τον εξή απλούστατο λόγο δεν σχεδιάστηκε ποτέ αυτός ο οργανισμός για τέτοιου είδου δουλειά, είδους δουλειά που καλείται τώρα να διεκπεραιώνει το 2016. Και έγινε και μια πρόσφατη έκθεση που ολοκληρώνεται αυτό το καιρό. Σε πολλούς τομεί είμαστε υποστελεχωμένοι Ουσιαστικά ένας άνθρωπος κάνει όλη τη δουλειά. Λοιπόν, δεν φτάνει αυτό. Χρειάζεται επιγόντως ενίσχυση σε επίπεδο προσωπικού για να παραμείνουμε, και να μπορούμε να διεκπεραιώνουμε όλο αυτό το φόρτο και να σα στέλνουμε όλα αυτά που μας ζητάτε ως νέες ευθύνες και υποχρεώσεις. Και προσβλέπουμε και υπολογίζουμε στο Κοινοβούλιο για να μας υποστηρίξει προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Ο κύριος Μέλο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πορτογαλικά αν δεν, με πειράζει, σας πειράζει. Δύο ερωτήσεις λοιπόν. Εγώ είμαι συγγετής στη Λίμπε για τη διαλειτουργικότητα και γι' αυτό ε, ζήτησα το λόγο και αξιοποιώ αυτό το τη που αναλογεί. Ο άλλο ε, έθεσε ερώτηση στην προηγούμενη συζήτηση. Λοιπόν, είναι ιστορική στιγμή που έχουμε μπροστά μας και θέλω να ρωτήσω το εξής. Η έλλειψη διαλειτουργικότητα διαλογικότητας έγινε περισσότερο αισθητή ιδίως με τα πρόσφατα γεγονότα στην Ευρώπη. Αλλά όχι μόνο το παράδειγμα των 14 ταυτοτήτων που εντοπίστηκαν στην περίπτωση της Γερμανίας είναι χαρακτηριστική. Θα μπορούσαν να αναφερθούν και άλλα παραδείγματα. Η δεύτερη ερώτηση που ήθελα να κάνω έχει να κάνει με το ποιες χώρες έχουν καταγράψει τις παλιότερες υποθέσεις με ανταλλαγή πληροφοριών, τέλος πάντων εκεί όπου η έλλειψη πληροφοριών φάνηκε ε, μοιραία. Δηλαδή, ξέρετε, χώρε στην Ευρώπη που ε, αντιστέκονται περισσότερο στην ανταλλαγή των πληροφοριών, που δεν συνεργάζονται αρκετά. Και αυτέ οι περιπτώσει έτυχε να υπάρξουν υποθέσει όπου είχαν μοιραίε επιπτώσει σε συγκεκριμένε χώρε. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να σα δώσω το λόγο. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Έχω την αίσθηση ότι δεν μπορώ να δώσω πλήρε απαντήσεις γιατί υπεύθυνοι για τέτοιου είδους δραστηριότητες θα είναι οι λειτουργικές υπηρεσίες και οι δύο προηγούμενοι ομιλητές από μένα θα μπορούσαν να σας δώσουν περισσότερα στοιχεία. Αλλά σε σχέση με τα, κοινά, τα κένα τα οποία υπάρχουν σε επίπεδο διαλειτουργικότητας είναι προφανή. Ένα άλλο παράδειγμα το είχαμε με τις επιθέσεις στο Παρίσι το 2015 είναι γνωστό σε όλους ότι ο ηγέτης αυτής της ομάδας είχε περάσει πολλές φορές τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε πάει πολλές φορές στη Συρία και αυτό δυστυχώς δεν καλύφθηκε και τελικά η έννοια της διαλειτουργικότητας αφ' αυτής είναι ένα τεχνικό μέσο το οποίο μόνο του δεν λύνει τα προβλήματα αλλά θα έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε σωστά. Ένα άλλο παράδειγμα το έχουμε στην απόκριση στην λεγόμενη μεταναστευτική κρίση. Παρακολούθησα αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές για την σχέση ανάμεσα στην παράνομη μετανάστευση και την τρομοκρατία. Υπήρχαν κάποιες εποχές ας πούμε στην Ελλάδα ε, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έφταναν εβδομαδιαία. Ε, δεν ήταν δυνατόν να τους ελέγξει κανείς με τον κατάλληλο τρόπο. Ακόμα και αν έγιναν λοιπόν οι έλεγχοι, τελικά παρόλα αυτά οι τρομοκράτες ίσως να μην είχαν δυσκολία για να μπουν στην Ευρώπη μέσα σε τόσο πολύ κόσμο. Αλλά η απάντηση περισσότερο στην ερώτησή σας ανήκει στις υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με τα θέματα αυτά στις χώρες μέλη. Τώρα για την ανταλλαγή ε, πληροφοριών. Η υπηρεσία μας δεν έχει εντολή να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο ανταλλάσσουν πληροφορίες τα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο μπορώ να πω όμως είναι ότι υπάρχει μια σαφή στάση αύξησης της χρήσης του ε, Σέγγεν. Όπως είπα ήδη από το 2016 είχαμε πάνω από 4 εκατομμύρια, από 4 εκατομμύρια έρευνες πολύ μεγαλύτερος αριθμός από το 2015 και για το 2017 πιστεύουμε αύξηση 25% στις έρευνες σε σχέση με το 2016. Συνεπώς το σύστημα ανταλλαγής ενημέρωσης και πληροφόρησης μέσω του Σέγγεν ως πλατφόρμα είναι κάτι το οποίο συνεχώς εξελίσσεται, αναπτύσσεται και εμπλουτίζεται. Υπάρχουν βέβαια κάποιες διαφορές στην συνεισφορά κάθε κράτους μέλους. Υπάρχουν μεγάλες χώρες που δίδουν πολλά στοιχεία και μικρότερες χώρες που δίνουν λιγότερα στοιχεία. Πάντως γενικά οι τάσεις νομίζω ότι είναι πλέον θετικές. Σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στη Μόνικα και μετά στην Κόμες. Σύντομες παρακαλώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Το θέμα είναι αν στον ενδιάμεσο χρόνο όλες οι χώρες μέλη έχουν δημιουργήσει τις απαραίτητες τεχνικές συνθήκες για να αξιοποιήσουν πλήρως ε, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, τι είδους υποστήριξη απαιτείται για να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Ευχαριστώ για την ταχύτητα και την αμεσότητα. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα συστήματα ανταποκρίνεται στις τεχνικές απαιτήσεις που υπάρχουν, αλλιώς δεν θα διασφαλίζαμε την, την ε, συνδεσιμότητα. Το θέμα δεν είναι όμως το τεχνικό κομμάτι, το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείται το προϊόν αυτή της διαδικασίας και γι' αυτό απαιτείται περισσότερη εκπαίδευση και κατάρτιση στα κράτη-μέλη για την χρήση του συστήματος αυτού. Νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι ο βασικός στόχος για την αύξηση της αποδοτικότητας και της ικανότητας να καλύψουμε τις τρομοκρατικές και εγκληματικές απειλές. Ήδη το σύστημα λοιπόν δουλεύει και αποδίδει, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ε, υποστηρίξουμε το σύστημα αυτό και να το βελτιώσουμε έτσι ώστε να λειτουργήσει πιο αποδοτικά και να πετύχουμε τους στόχους τους οποίους έχουμε. Έχουμε μέσα τα οποία είναι λειτουργικά και θα έλθουν και καινούρια μέσα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Η Άννα Γκόμες. Ευχαριστώ κύριε Γκαρκόφ. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Έχετε ασχοληθεί με το θέμα της ακεραιότητας και της λειτουργικότητας των τραπεζών δεδομένων τις οποίες διαχειρίζεστε. Να το πω αλλιώς, εσείς ή κάποιοι άλλοι ίσως έχουν κάνει μια ανάλυση ποιοτική των στοιχείων. Υπάρχουν πολλά στοιχεία σαν παράδειγμα για τους ετούντες άσυλο, για τους μετανάστες κτλ αλλά τι γίνεται με κάποια εθνικά προγράμματα όπως οι λεγόμενες χρυσές βίζες, χρυσές θεωρήσεις όπου οι πολύ πλούσιοι από τρίτες χώρες αγοράζουν ουσιαστικά την εθνικότητα ή την υπηκότητα μάλλον. Ε, και φυσικά υποτίθεται ότι πρέπει να έχουν καθαρό ποινικό μητρό, αλλά στις χώρες από τις οποίες προέρχονται είναι εύκολο να αγοράσουν ένα καθαρό ποινικό μητρό. Συνεπώς λοιπόν τι δεδομένα έχετε και σε ποιο βαθμό συνδέεται με τις θεωρήσεις για το Σέγγεν αυτή η διαδικασία. Ιδιαίτερα για κάποια προγράμματα Ευχαριστώ για την ερώτησή σας κυρία Γκόμες. Ε, ο οργανισμός μας είναι αρμόδιος και με μεγάλη σοβαρότητα ελέγχει πραγματικά την ποιότητα των δεδομένων στο κεντρικό σύστημα. Κάνουμε ελέγχους ε, και στέλνουμε και εκθέσεις ποιότητας στα κράτη-μέλη όταν βλέπουμε παρατυπίες, προβλήματα ε, με τα δεδομένα και μετά είναι ευθύνη των κρατών μελών να τα διορθώσουν. Έτσι είναι η κατανομή των αρμοδιοτήτων. Εμείς σε το σύστημα λειτουργούμε και ε, χειριζόμαστε, δεν έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα η απάντηση ε, στο δεύτερο είναι όχι. Δεν έχουμε ούτε εντολή ούτε αρμοδιότητα να ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Τα κράτη-μέλη είτε μεμονωμένα είτε συνολικά, συλλογικά ασχολούνται με τα δεδομένα και για αυτό που λέτε για τις θεωρήσεις. Αλλά εμείς εγγυόμαστε ότι όλα τα συστήματα ε, που διαθέτουν τα κράτη-μέλη να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους είναι σωστά και να ελέγξουν αν κάποιος έχει ποινικό μητρό ή εκκρεμούν εις βάρου κάποιες διαδικασίες ή ακόμα έχει ζητήσει και αλλού θεώρηση και του έχει ε, κάποια αρχή αρνηθεί την έκδοση αυτής. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιούν τις δυνατότητες του συστήματος στα κράτη-μέλη ο δικός μας οργανισμός έχει τεράστιες δυνατότητες και ευκαιρίες αν ενισχυθεί με τις απαραίτητες ε, υπηρεσίες και τους πόρους για να κάνει περισσότερα και να βελτιώσει και τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη για να μπορούν εκείνα με τη σειρά τους να τα ε, αξιοποιούν. Η κυρία Γκόμες επανέρχεται. Αν δείτε, ας πούμε, ότι ένα κάποιο κράτος μέλος ξαφνικά εκδίδει πολύ περισσότερες θεωρήσεις από ό,τι προηγουμένως ή κανονικά για πολίτες μιας συγκεκριμένης χώρας. Αυτό χτυπάει κανένα καμπανάκι ε, στις ε, υπηρεσίες. Ε, ε, εσείς ενημερώνετε καμία αρχή. Ξαφνικά, ας πούμε, υποθετική περίπτωση, ε, βίζες για Σέγγεν ε, ε, από τη Μάλτα σε πολίτες ας πούμε Λίβιους. Αυτό χτυπάει κανένα καμπανάκι σε εσά, ε, σας ανησυχεί. Κατανοώ την ερώτηση, ναι. Εμείς δίνουμε στατιστικές εκθέσεις, εκδίδουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα και στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε μια τέτοια περίπτωση, τέτοιου είδους, ότι ας πούμε αυξάνονται οι βίζες Σέγγεν για κάποιο διάστημα, βεβαίως το ανοιχνεύουμε και το αναφέρουμε. Τώρα τι δράση θα αναλάβουν τα κράτη-μέλη δική τους υπόθεση ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν υπάρχει ανάγκη νομοθετικής πρωτοβουλίας ή άλλη συνέχεια που δίδεται. Βεβαίως το πρότουμε αυτό εμείς ε, τακτικά στις εκθέσεις μας. Ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρον και πολύ συγκεκριμένο αυτό. Τελευταίος εγγεγραμμένος ο μιλητής, ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρ. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Δεν λειτουργούν τα μικρόφωνα. Α, εντάξει τώρα. έχει να κάνει και με ερωτήσεις που έχω κάνει στους προλαλήσαντες στο προηγούμενο πάνελ. Υπάρχουν διαφορετικά... Έκλεισε το μικρόφωνο το μιλητή. Ε, ξέρουμε ότι η υπηρεσία σας είναι ουδέτερη σε σχέση με τις διάφορες συνταγματικές ε, καταστάσεις στα κράτη-μέλη. Αλλά επειδή επιμένετε ότι η αποστολή σας είναι να εξασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων ε, και να ελέγχετε την ποιότητα και την αξιοπιστία τους, έχετε μέχρι τώρα εμπειρία ως προς την εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων, ε, αστυνομία, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπηρεσίες Πληροφοριών. Τα ίδια στοιχεία και δεδομένα ισχύουν και με τον, με τον ίδιο τρόπο τα υποβάλλουν όλες οι χώρες, είτε είναι το Βέλιο, είτε είναι η Γαλλία κτλ. Ναι. Καλά, ποτέ δύο χώρες δεν κάνουν ακριβώς τα ίδια. Υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα, αλλά ειλικρινά δεν έχω μελετήσει τις διαφορές από το πρίσμα αυτό που το βλέπετε εσείς, αλλά από την εμπειρία μου, δεν συνδέεται αυτό απαραίτητα με τα δεδομένα, αλλά θα έλεγα λοιπόν εκ πείρας ότι ο συντονισμός του έργου μεταξύ του οργανισμού και των ε, χωρών που έχουν συγκεκριμένες συνταγματικές επιταγές είναι πιο δύσκολο από ότι να μην υπάρχει αυτό στα συντάγματα των χωρών. Merci. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, ούτε ζητεί κανείς άλλο το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ποιοτική αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Ίσως συντομεύτηκε κάποιος γιατί πολλοί συνάδελφοι έχουν πάει στην Ολομέλεια γιατί ψηφίζουμε σε λίγο σε ένα τέταρτο και είχαν μάλλον άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις ε, για τους καταλόγους ψηφοφορίας. Πάντως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την άμεση και ειλικρινέστατη, όσο και ακριβέστατη ανταλλαγή απόψεων. Ε, πολλές προφορίες μας δώσατε, ε, ακριβώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τις δύο συνεισηγήτρες, τη Χέλγκα Στέβενς και την Μόνικα Χόλμαϊερ. Ευχαριστούμε πολύ και για τις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις των συναδέλφων για να καταλάβουμε τι γίνεται και να χαράξουμε και τις προοπτικές για το μέλλον που να είναι πραγματικά θετικές και χρήσιμες. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γκάρκοφ. Ε, ελήφθηκε το μήνυμα πάρα πολύ <laughs> καλά ότι έχετε περισσότερες ανάγκες για να αντιμετωπίσετε την απειλή που είναι τόσο σημαντική και θα πρέπει τα κρατημέλη να το καταλάβουν γιατί ανατρέχουν όλο και περισσότερο στην υπηρεσία σας. Ε, έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ε, χρήση των κρατών μελών, των υπηρεσιών σας. Ε, έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι πολύ σημαντικές. Ευχαριστώ που ήρθατε να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που δεχτήκατε αυτούς τους κανόνες που ήταν έτσι λίγο αυστηροί και σφιχτοί ε, αλλά είναι πινκ-πονγκ αυτό ερωταπόκριση και δεν είναι καθόλου εύκολο να απαντάει κανείς. Ευχαριστώ πολύ, καλές ψηφοφορίες, καλή σας μέρα και καλή επάνωδο.